επιβεβαιώνεται αυτός ο διορισμός. Τετάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού θα υπογράψω δύο ε, νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία και οι τίτλοι θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στην έγκριση